Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη από όλους σας. Και πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπιανκόφσκα, την κυρία Επίτροπο που άργησα, αλλά και οι δύο ήμασταν σε συνεντεύξει τύπου κάτω. Και μετά τη συνέντευξη τύπου οι δημοσιογράφοι ρώτησαν και κάποιες ρωτήσαν την κυρία, την κυρία Μπιανκόφσκα και μετά θέλω να απαντήσω κι εγώ. και τουλάχιστον έπρεπε να περάσω 7 λεπτά με δημοσιογράφους για να συζητήσουμε το διάφορα προβλήματα, να συζητάμε τα προβλήματα με τους δημοσιογράφους είναι πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές μας. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν ξανά κυρία μου και από εσά ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχετε την ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως, την έχετε μπροστά σας. Επιθυμείτε κάποια αλλαγή? Έχετε κάποια σοβαρή αλλαγή να προτείνετε. Μην διστάζετε. Δεν βλέπω να σηκώνετε χέρι. Οπότε είστε κατά των αλλαγών. Εγώ δεν έχω ανακοινώσει του Προέδρου. Αυτά είναι υπέροχα μαντάτα για όλους. Και ξεκινάμε το σημείο εμείς της διάταξης. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του ματολογίου του Ευρωπαϊκού για τη βιομηχανία, ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Σβέθα Μιακόψια που είναι υπεύθυνη για την εσωτερική αγορά, τις, μικρομεσ... τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Συνάντησα περίπου 15 μέλη τη επιτροπή μας, συναντήσαμε την κυρία Μπιανκόφσκα την περασμένη εβδομάδα, συζητήσαμε ε, την αμυντική βιομηχανία, σημαντικότατο θέμα, Είχαμε 19-20 ευρωβουλευτές από την ΙΜΚΟ, την ΤΕΒΕ, όχι την ΤΕΒΕ, ΣΕΝΤΕ, ΙΜΚΟ, ΣΕΝΤΕ και ΉΤΡΕ. Και 15, τα 2 τρίτα αυτών, 3 τέταρτα αυτών, ήταν μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ, διότι ενδιαφερόμαστε πολύ για την βιομηχανική πολιτική. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, κυρία Επίτροπε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ότι θα θέλατε να μας ενημερώσετε ίδια για το περιεχόμενο της Επιτροπής, της επιστολής συγγνώμη, που στείλατε προς τους Υπουργούς. Είδαμε την επιστολή και αυτό που είναι σημαντικό είναι να βοηθήσουμε ε, τη βιομηχανία μας και θέλετε να ολοκληρωθεί και ο τριμερής διάλογος για την ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών. Πιθανότατα θα ήταν δυνατόν την επόμενη εβδομάδα τη Δευτέρα από πλευράς της Επιτροπής μας η κυρία Πιλάρντε Καστίγιο Βέρα είναι η βασική διαπραγματεύτρια και εγώ είμαι υπεύθυνο σαν πρόεδρος της Ήτρε για τον τριμερή διάλογο και ε, να οδηγήσω το διάλογο αυτό σε επιτυχία. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, έχετε το λόγο και θα θέλαμε να κάνετε την αρχική σας παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Αισθάνθηκα ότι ήταν σημαντικό να συναντηθώ μαζί σας το ταχύτερο δυνατό για να σας εξηγήσω την επιστολή που απέστειλα στο Συμβούλιο στους 28 υπουργούς, υπουργούς για την νέα προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε για την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Είναι και μια ευκαιρία για σας να θέσετε ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Είναι ένα αρχικό έγγραφο αυτό που αναφερόμαστε στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, αλλά είναι σημαντικό βήμα. Η προσέγγιση είναι αρκετά νέα, γι' αυτό ήταν και σημαντικό για μένα να μοιραστώ τις απόψεις μαζί σας. Θεώρησα ότι θα ήταν χρήσιμο να σας θέσω το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τι σημαίνει στην πράξη η προσέγγιση μας και πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πω ότι η βιομηχανία είναι στο επίκεντρο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιπροσωπεύει 35 εκατομμύρια θέσεις εργασία και πάνω από τις μισές εξαγωγές χρηματοδοτεί 80% της ιδιωτικής έρευνας και ανάπτυξης και βέβαια συμβάλλει κατά σημαντικό τρόπο στις, στα οικονομικά κέρδη λόγω παραγωγικότητα. Αλλά θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από κληρονομιά. Θέλουμε να δημορφώσουμε και το μέλλον τη, Θέλουμε ισχυρή, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θέλουμε να παράγει θέσει εργασία τώρα και στι επόμενε δεκαετίε, Και γι' αυτό ε, έχουμε ετοιμάσει μια στέρεη βιομηχανική βάση και τη θεωρούμε προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, μηχανολογία, στην αεροναυπηγική, στη χημική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία εγούμεθα. Αλλά ίσω σε άλλου ε, τομεί θα μπορούσαμε να επαναβιομηχανοποιήσουμε την Ευρώπη. Έχουμε επιχειρήσει που συνεχώ είναι στην αιχμή τη καινοτομία, τη έρευνα και τη ανάπτυξη Τρία τέταρτα των ε, ε, επιχειρήσεων έχουν εισαγάγει καινοτομίε τα τελευταία τρία χρόνια. Αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα για προκλήσει. Το ξέρετε καλύτερα από εμά. Έχουμε ένα κενό επενδυτικό 400 δισεκατομμύριων ευρώ όσον αφορά την παραγωγικότητα και η οικονομική κρίση έχει πλήξει την βιομηχανικό τομέα για πολλούς λόγους, ιδιαίτερα σκληρά. Μειώθηκε πάνω από 9% από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι τον Ιανουάριο 2014. Το 2000 το 2014 η απασχόληση στην κατασκευή και στην βιομηχανία μειώθηκε στον κάτι μέλη εκτός μίας. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 6% αλλά στην Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία μειώθηκε ε, περισσότερο από 30% και όπως βλέπουμε τώρα, η οικονομική μας ανάκαμψη, η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη είναι πολύ πιο αργή από τις άλλα μέρη του κόσμου, διότι η παραγωγή στην Ευρώπη το 2014 ήταν ακόμα 9% χαμηλότερη από την ακμή της το 2008. Σε κάποιους βασικούς τομείς ε, είμαστε πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Πράγματος χάρη δεν επενδύουμε αρκετά σε νέες τεχνολογίες το ποσό που επενδύθηκε από τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και συμπενθυμίζω 8% αυτού ε, γίνεται στη βιομηχανία, στους βιομηχανικούς τομείς, είναι μόνο 40% του ποσού που επενδύεται στις ΗΠΑ. Μία νέα έρευνα δείχνει ότι περίπου το μισό από τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν έχουν χρησιμοποιήσει προωθημένες βιομηχανικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε σχεδιάζουν να κάνουν κάτι τέτοιο τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι μια νεα ερευνα δειχνει οτι περιπου το μισο απο τις επιχειρησεις ευρωπαικης ενωσεω δεν εχουν χρησιμοποιησει προθυμένε βιομηχανικες τεχνολογιες στην ευρωπαικη ενωση ουτε σχεδιαζουν να κανουν κατι τετοιο τα επομενα χρονια αυτο ειναι μια προκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ακόμα εκεί που ηγούμεθα παραδοσιακά αισθανόμαστε πάρα πολύ ισχυρές ανταγωνιστικέ πιέσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι μόνο η τέταρτη περιοχή στον κόσμο όσον αφορά την καινοτομία, πίσω από την Νότια Κορέα, τι Πολιτείες και την Ιαπωνία. Παραδείγματο χάρη, στον τομέα των χημικών η Ευρώπη χάνει το πλονέκτημά τη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ λόγω της εκμετάλλευσης του αερίου σχιστολίθου από τις αμερικανικές εταιρείες. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι παραπάνω από στατιστικά στοιχεία. Αυτό αφορά και την έλλειψη ευελιξίας πραγματος χάρη. Μπορώ να σας δώσω ε, λίγα λόγια για πρόσφατη συνάντησή μου και ανησυχητικό παράδειγμα αποτελεί τις προάλλες συνάντησα. Μια πολύ μεγάλη πολυεθνική με σημαντικές επιχειρήσεις όλο τον κόσμο μου είπε ότι είχε ένα πρόγραμμα για το οποίο θα προσελάμβανε 500 ε, μηχανικούς με ψηλά προϊόντα, ε, προσόντα και ερευνητές για τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Και βέβαια ε, λειτουργεί σε ευρύ πλαίσιο σε πολλά δυτικά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Θα μπορούσε να έχει βρει προσωπικό με τα αναγκαία προσόντα σε αυτό το κράτος μέλος και θα προτιμούσε να προχωρούσε σε εκείνη τη χώρα αλλά τελικά αποφάσισε ότι δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τους ε, κινδύνους και ήθελε να κατασκευάσει την εγκατάσταση εκτός Ευρώπης. Γιατί? Διότι αν μετά από δύο-τρία χρόνια ακμής η επιχείρηση δεν χρειαζόταν όλα αυτά τα άτομα, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί ιδεόντως. Λοιπόν, 500 θέσει εργασία προστιθέμενη αξία υψηλή ε, για τουλάχιστον 2-3 χρόνια χαθήκαν την Ευρώπη. Ποιο κέρδισε στην Ευρώπη από αυτό, θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να είμαστε συνετοί και σοφοί όσον αφορά τη λύση που θα βρούμε. Σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πρακτικά σωστή προσέγγιση. Υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται ότι θεωρούν ότι η λύση είναι να κλείσουμε την πόρτα στου ξένου ανταγωνιστέ ή να επιβάλλουμε περαιτέρω απαιτήσει. Βέβαια προσπαθώ να καταλάβω αυτή την άποψη, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αυτό που κάνει είναι να μειώνει την επιλογή και να αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Η λύση είναι να αυξήσουμε εμείς αυτά που προσφέρουμε, να δώσουμε πλαίσιο στήριξη στι επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν και θέλουμε μια ανοιχτή και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη βιομηχανία. Λοιπόν, τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκολύνουμε τις εταιρείε να εντάσσονται στην ενιαία αγορά και στις παγκόσμιες, στα παγκόσμια κυκλώματα και πρέπει να ετοιμάσουμε ε, τα σωστά δίκτυα, έτσι λειτουργεί ο κόσμο με αυτά τα δίκτυα δεν υπάρχει κανένα προϊόν που, σχεδόν που να έχει κατασκευαστεί μόνο από μία επιχείρηση. One Δεν υπάρχει κάτι που κατασκευάζεται από μία εταιρεία σε ένα εργοστάσιο, σε ένα μέρος και να κάνει την έρευνα, το σχεδιασμό και την παραγωγή και το προϊόν να ξεκινά και να τελειώνει σε μία εγκατάσταση. Διάφορα τμήματα του προϊόντος αναπτύσσονται από διαφορετικές εταιρείες σε διαφορετικούς τομείς, διαφορετικά γραφεία σε όλο τον κόσμο και εγκαταστάσεις. Λοιπόν, οι πιο επιτυχείς μας εταιρείες εργάζονται μέσα σε μια λυσίδα συνεχή, ψηφιακή τεχνολογία. Έχουμε διάκριση μεταξύ υπηρεσιών και ε, κατασκευής και παραγωγής που είναι όλο και πιο μικρή η διάκριση. Αποτελούν μια ενότητα. Χρειάζονται ριζοσπαστικές λοιπόν αλλαγές που ήδη λαμβάνουν χώρα. Πρώτα απ' όλα η ψηφιοποίηση επιτρέπει στους κατασκευαστές να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των διαφόρων πελατών χωρίς να χάνουν το πλεονέκτημα της παραγωγής κλίμακας είναι μαζική παραγωγή σύμφωνα με τον κάθε πελάτη. Μετά για τις εταιρείες είναι πιο εύκολο και πιο επικερδές να αμαδοποιούν αγαθά και υπηρεσίες μαζί. Και τρίτον, αυτό επηρεάζει όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα προϊόντα θα προσφέρονται σαν ένα. Το παραγόμενο αγαθό και συνοδευόμενες ε, ε, υπηρεσίες. Το αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, θα γίνεται ένα πιο ε, εξατομικευμένο προϊόν, μοναδικό προϊόν, ε, ε, πέρα από αυτό, οι αυτοκινητομηχανίες όχι μόνο πουλούν τα αυτοκίνητά τους, αλλά προσφέρουν και μεταπόληση υπηρεσίες, συντήρηση ή ασφάλεια. Ε, ίσως να αλλάξει η δουλειά του κατασκευαστού αυτοκινήτου από το να πουλά απλώς ένα αυτοκίνητο μέχρι να πουλά τώρα να γίνει το να πουλά υπηρεσίες κινητικότητας. Θα επιτρέψει αυτό στις εταιρείε να εκμεταλλευτούν την προστιθέμενη αξία σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής και προσφοράς δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε σε ένα κομμάτι της αλυσίας αυτής της εταιρεία. Θέλουμε να ηγούνται εταιρείε μας στους τομείς που δίνουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, επειδή αγαθά και υπηρεσίες γίνονται τόσο αλληλένδετα πράγματα, οι περιορισμοί στις υπηρεσίες, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα πλήξουν την πώληση των αγαθών. Άρα θα πρέπει να έρθουν τα βασικά εμπόδια και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην ενιαία μας αγορά. Το δεύτερο τμήμα τη νέα βιομηχανική μα προσεγγίσεω είναι να προωθήσουμε τον εξυγχρονισμό τη βιομηχανία Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τι εταιρείε Ευρωπαϊκή Ένωσης να προσαρμοστούν δεόντως είτε μέσω ψηφιοποίησεω είτε μέσω αναπτύξεω τεχνολογιών αποδοτικών στον αφορά την ενέργεια ή να έχουμε τεχνολογίε εχμής που θα αναπτύξουμε. Για μία ακόμη φορά έχουμε πολλέ ευρωπαϊκέ εταιρείε που ήδη είναι επιτυχεί. Να σας ε, δώσω ένα παράδειγμα ψηφίσεως. Την περασμένη ε, εβδομάδα είδα τι έκανε μια εταιρεία ε, που ασχολείται με μεγάλο όγκο στοιχείων και την ασφάλειά τους. Είναι πολύ σημαντικό θέμα κατεπήγον. Σύμφωνα λοιπόν με τη βιομηχανία αυτή η εταιρεία παρέχει τεχνικές λύσεις για να προστατεύσει βιομηχανικά στοιχεία για να μην έχουν πρόσβαση τα μέρη σε αυτά τα στοιχεία, να είναι εμπιστευτικά και αυτή είναι μόνο μια ευρωπαϊκή εταιρεία που ανταγωνίζεται με τέσσερις αμερικανικές ανταγωνίσεις εταιρείες στον κόσμο. Χρειαζόμαστε περισσότερες εταιρείες σαν και αυτή, την ευρωπαϊκή, αλλά αυτό που χρειάζονται αυτές οι εταιρείες είναι σαφείς κανόνες για την χρήση των ογκωδών ε, δεδομένων και να επιτρέπεται η ανοιχτή πρόσβαση, δηλαδή εργατικό δυναμικό με τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις. Όλες οι εταιρείες όταν κουβεντιάζουν μαζί μου μου λένε ότι κατεπηγόντως το χρειάζεται αυτό. Τώρα το 1 πέμπτο των ε, αποφύτων των πανεπιστημίων εργάζονται σε μέσα και χαμηλά επίπεδα στον δεξιότητε και αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη. Χρειάζεται να είναι έτοιμο το εργατικό δυναμικό για την ψηφιακή εποχή. Υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη επαγγελματιών στον ψηφιακό τομέα και αυτή θα πρέπει να καλυφθεί. Θα ξέρετε ότι φέτο θα, θα υπάρχουν πάρα πολλά κενά στον τομέα ε, τον ψηφιακό και αυξάνεται, αυξάνονται οι ανάγκε στηρίζω και τη μεταποίηση, τη μετατροπή του ψηφιακού τομέα. Πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των ενεργειακών μας πηγών. Η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βασική αρχή της Ενεργειακής Ένωσης ε, που υποστηρίζω ένθερμα. Η ενεργειακή απόδοση σημαίνει και χαμηλότερες εκπομπές. Θα πρέπει να έχουμε μικρότερη ε, μόλυνση, να είμαστε πιο αποδοτικοί οικονομικά και χρειάζεται και συνεργασία με το βιομηχανικό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι είναι προβλέψιμο και είναι κάτι που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Θέλουν να ξέρουν τι θα γίνει σε 5, 10, 15, 20 χρόνια στην Ευρώπη η βιομηχανία. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ ανταγωνιστική βιομηχανία και βιομηχανία που ανταποκρίνεται στι ανάγκε για την ενέργεια και για το κλίμα. Και επίση θα πρέπει να ηγηθούμε των συζητήσεων σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία όσον αφορά αυτά τα θέματα που προανέφερα. Και τέλος χρειαζόμαστε ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Θα πρέπει το ενεργειακό μείγμα το διαφυλάξουμε. Δεν είναι μόνο σημαντικό για τη βιομηχανία μας, αλλά πρωτίστως για την ασφάλειά μας. Εάν θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει σημαντικό φορέα και παίκτη στο παγκόσμιο προσκήνιο, πρέπει να είναι καινοτόμα βιομηχανία και να δημιουργήσει πιο προθυμένε τεχνολογίε. Α πάρουμε ένα παράδειγμα. Δύο τομεί όπου η Ευρώπη είναι στην πρώτη γραμμή τη τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία. Είναι η άμυνα και το διάστημα. Μόνο δύο φράσει να πω γι' αυτό. Διότι, όπω είπα πριν, είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με εκπροσώπου τη αμυντική βιομηχανία την περασμένη εβδομάδα. Όσον αφορά το διάστημα, η Ευρώπη μέσα των δύο βρασικών προγραμμάτων Κοπέρνικος και Γαλιλαίος αναπτύσσει ε, πολύ ανταγωνιστική και πολύ καινοτόμα βιομηχανία και όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία βλέπουμε δραματική μείωση των ερευνητικών δαπανών και στην αμυντική βιομηχανία. Χρειαζόμαστε ισχυρή αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη που επενδύει στην έρευνα και που εξακολουθεί να ηγείται στην καινοτομία και θα πρέπει να ωφελείται πλήρως από την ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά. Λοιπόν, το τρίτο τμήμα τη Νέα προσέγγιση είναι να εξασφαλίζουμε ότι είναι φιλικό το περιβάλλον για τι επιχειρήσει. Αυτό είναι ο ευρύτερο ε, τομέα που πρέπει να εξετάσουμε, διότι οι ευφυεί τεχνολογίε πραγματικά χρειάζονται και ευφυέ βιομηχανικό κλίμα. Πριν από κάποιου μήνε. Κάποιο διευθύνων σύμβουλο ε, μια εταιρεία που παράγει ιατρικέ συσκευέ μα είπε ότι η ενιαία αγορά έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να επεκταθεί διασυνοριακά αλλά για τη δανειοδότηση, για τη δανειοληψία έπρεπε να προσφύγει στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά αυτό αφορά και την καλύτερη νομοθεσία, λιγότερες ρυθμίσεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος τον κάθε τομέα και τι ανάγκες έχει. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πετύχουμε τα στοιχεία, τους στόχους που θέλουμε. Πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να βρούμε ποιες είναι ευκαιρίες που υπάρχουν για ανάπτυξη και γι' αυτό σαν απομονω... εκτός απομονωμένη ε, στρατηγική θα πρέπει μάλλον την αγωνιστικότητα τη μηχανική να βάλουμε στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα πρέπει να σαμώνται σε όλες τις πολιτικές. Όλες οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει αυτή την απόχρωση τη βιομηχανική. Το σημάδι των βιομηχανικών το έχουν όσοι πολιτικές. Σε κάθε στρατηγική που θεσπίζουμε. Στατική Ενεργειακή Ένωση, για την Κεφαλουχική Ένωση κλπ. Ψηφιακή Ένωση, ενιαία αγορά. Μέχρι το τέλος του έτους για τη στατική αυτή χρειαζόμαστε στρατηγική που προωθεί τι επενδύσει, που προωθεί την καινοτομία, στρατηγική που βοηθά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τι νεοφύει επιχειρήσει και στρατηγική που πραγματικά δεν λησμονεί του καταναλωτέ. Χωρί καταναλωτέ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει αγορά. Μετά θα πρέπει να έχουμε μια ε, σωστή προσέγγιση, να χρησιμοποιούμε σωστά τους πόρους με αποτελεσματικό τρόπο, Πρέπει να βελτιστοποιούμε τη χρήση αυτών. Η νομοθεσία μας θα πρέπει να λειτουργεί μέσω καλύτερης επιβολής και υλοποίησης, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό. Θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και γι' αυτό διοργανώνουμε ε, μια αλλαγή νοτροπίας αντί από ξεχωρισμένες δράσεις και σχέδια δράσεων για το χάλιβα, για τη φαρμακοβιομηχανία κλπ. Έχουμε ενιαία ολοκληρωμένη προσέγγιση και σχέδιο, εξετάζοντας βέβαια την ιδιαιτερότητα κάθε τομέα. Και τρίτον, θα πρέπει να εργαστούμε σε συμπράξεις και εταιρικέ σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρήσεων και εγώ συνεχώς ακούω τι μου λένε και τι ανάγκες έχουν. Είμαι Οκτώ μήνες τώρα ακούω. Ακούω τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες, τις εταιρείες, τους καταναλωτές. Αφού γκράζομαι τις απόψεις τους. Θέλουμε συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών, διότι πολλές ευθύνες, μεγάλη ευθύνη για τη βιομηχανία είναι στους δικούς, τους, ε, δικούς τους Και τέλος, χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εξού και η παρουσία μου εδώ σήμερα, κοινό ρόλο είναι να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε συνθήκε ώστε οι επιχειρήσει να χρησιμοποιήσουν το υπάρχον δυναμικό, τι δυνατότητε που έχουμε. Θέλουμε βέβαια τη χρήση των εργαλείων τη ενιαία αγορά για να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό προστατεύοντα του καταναλωτέ και παραμένοντα ανοιχτοί στον κόσμο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει η βιομηχανία, θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη βιομηχανία χρειάζεται να έχουμε ισχυρή ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας για αυτή την ομιλία που αποτελεί και την αρχή των συζητήσεών μας για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Βιομηχανία, την Ανάπτυξη και την Εφαρμογή. Θα ξεκινήσει η συζήτηση τώρα με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων καταρχάς και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Νίμπλερ να λάβει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Κυρία Νίμπλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω θερμά την ε, κυρία Επίτροπο για το ότι ήρθε σήμερα για αυτήν την αλληλεγγυη απόψεων στην Επιτροπή μα. Και καταρχά μία διαπίστωση. Θεωρώ αξιέπαινο το γεγονό ότι η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Μα είπατε ξεκάθαρα πώ χρειάζεται η δημιουργία και η σύσφυξη των ε, εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στι επιχειρήσει, στη βιομηχανία και στην ε, πολιτική και φυσικά ε, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε ανταγωνιστικοί και ε, σε αυτό ε, περιλαμβάνεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας η βιομηχανία δεν είναι μόνο σημαντική σε διεθνέ επίπεδο, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι έχετε πάρει την απόφαση με ξεκάθαρε και συγκεκριμένε προτάσει να στηρίξετε την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχουν σίγουρα λεπτομέρειε οι οποίε χρειάζονται επεξεργασία και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε λεπτομέρειες του προγράμματος REFIT για παράδειγμα, τις καλύτερες νομοθεσίες, την περαιτέρω εξέλιξη της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Πάρα πολλά ερωτήματα λοιπόν ε, μας απασχολούν σε αυτούς τους ε, τομείς. Επίσης γίνεται λόγος για την βιομηχανία 4,0 ε, και το τι χρειαζόμαστε σε πολιτικό πλαίσιο, σε νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τις ε, μεσαίες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ψηφιακά και εμεί. Θα ήθελα λοιπόν να επεκταθείτε λίγο σε αυτό, να μας πείτε πώς ακριβώς ε, σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις ή κάποιες ιδέες. Να πω επίσης πως με πολύ χαρά άκουσα τα σχέδιά σας για την ε, στρατηγική για την εσωτερική αγορά, η οποία θα ε, διασυνδέεται και με την ε, παγκόσμια βιομηχανία. Τώρα, μία ερώτηση που εμπίπτει στις δικές σας αρμοδιότητες δεν αναφερθήκατε σήμερα στην εναέρια κυκλοφορία, στους δορυφόρους και στην αεροπλοεία, κάτι που θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δύο ε, προγράμματα, ο Κοπέρνικος και το πρόγραμμα Γαλιλαίος, τα οποία ε, είχαν αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες ε, στην εφαρμογή του στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, είναι οι εξελίξεις, τι γίνεται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να εξελίξετε τα προγράμματα αυτά, τι σκοπεύετε να κάνετε τα, τα επόμενα πέντε χρόνια, εάν υπάρχουν προτάσεις για νέα διαστημικά προγράμματα, αν τα, προγράμματα, τα εφιστάμενα προγράμματα έχουν ε, εξελιχθεί η διαστημική πολιτική μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή Ήτρε και ιδιαίτερα ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος των κρατών μελών και το πώς ε, αυτά συνδέονται με την περαιτέρω βιομηχανική εξέλιξη της Ευρώπης. Έχετε κάποιες ε, προτάσεις ιδιαίτερα για το πώς μπορούμε να επεκτείνουμε να εξελιχθούμε στον τομέα αυτό και τι γίνεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Έπειτα, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν προτάσεις για νέα χρηματοδοτικά μοντέλα για τα προγράμματα Γαλιλαίος και Κοπέρνικος. Στην, ε, στο τελευταίο συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ε, διάστημα, Ακούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τι ε, σκοπεύει να κάνει η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ποιε είναι οι νέε δομέ που δημιουργούνται έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τα διαστημιακά του προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πλευρά ε, τέτοιε ανάλογε ή αντίστοιχε τέλο πάντων προτάσει. Αυτά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων και αναμένω την απάντησή σα με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κάθε συντονιστής έχει τέσσερα λεπτά να σας υπενθυμίσω. Ε, τα ξεπεράσατε. Κύριο Μαρτέλ, τώρα εκ μέρους των ε, Σοσιαλδημοκρατών, έχετε την δυνατότητα να μιλήσετε για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω πάνω από μισή λεπτά. Παρακολούθησα τις ε, διαπιστώσεις της ε, Επιτρόπου και μπορώ να συμφωνήσω με πολλά πράγματα για τις διαπιστώσεις που κάνει. Δυστυχώς ε, θα ήθελα να είχαμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπατε και εσείς, για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για τις επενδύσεις, πού υπάρχουν προβλήματα. Σίγουρα η ευρωπαϊκή ανάκαμψη είναι σημαντική, αλλά οι επενδύσεις αποτελούν και το ευάλωτο σημείο μας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν συμφωνείτε να επανεξετάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον ορισμό των ε, ε, σχετικών αγορών ε, πολλές φορές είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό, ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος ε, και εμείς έχουμε συστήματα τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 80 και δεν είμαστε καθόλου εξυγχρονισμένοι. Ε, μία μεγάλη πολυεθνική, για παράδειγμα, ένας γίγαντας όπως η Airbus, ε, η Airbus δεν μπορεί να ε, ανταπεξέλθει και χρεοκοπεί και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Θα ήθελα επίσης να δούμε αν υπάρχουν πολιτικές για να μπορέσουμε να έχουμε ισότιμα ουσόρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο στην Ευρώπη, διότι υπάρχουν αποκλήσεις και σε εσωτερικό επίπεδο. Επίσης αναφερθήκατε στην έλλειψη ευελιξία στην Ευρώπη και αυτό πραγματικά με προβληματίζει λίγο, διότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα κοινωνικά μας μοντέλα. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη τα δικαιώματα των εργαζομένων σήμερα σχετίζονται με τις συμβάσεις εργασίας. Εάν θέλουμε να είναι λίγο πιο καθησυχασμένοι οι εργαζόμενοι όταν εργάζονται σε επιχειρήσεις ε, ε, χρειάζονται και εγγύησεις που να αφορούν τους εργαζομένους και όχι μόνο τη συμβάση εργασίας. Αυτό αποτελεί πρόβλημα και πρέπει να ανακτηθεί εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας. Ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και κάποια χρόνια. Το κεφάλαιο δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει κινδύνους και ε, οι κίνδυνοι ε, διαχέονται στους εργαζομένους και το σχέδιο Juncker να υπενθυμίσω ότι θέλει απλώς να καθησυχάσει τις αγορές, να καθησυχάσει τους επενδυτές για να τους πει ορίστε, ελάτε σε εμά, ακόμα και αν έχετε πρόβλημα να λαμβάνουμε εμεί τους κινδύνους για αύριο και επομένω πρέπει να τα επανεξετάσουμε όλα αυτά. Και επίση θα πρέπει να πω ότι τι είναι επιχείρηση. Αναφερθήκατε σε επιχειρήσει και συμφωνώ και εγώ μαζί σα. Η επιχειρήση είναι κεφάλαιο, αλλά αποτελείται από άνδρε και γυναίκε. Και εδώ πραγματικά θα ήλπιζα να μας πείτε και την άποψή σας για τον κοινωνικό διάλογο, που είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πλούτο στις κοινωνίες μας. Και επίσης, βλέπουμε πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις που σήμερα μπορούν να ανταπεξέλθουν ενώπιον του παγκόσμιου ανταγωνισμού είναι οι, χώρες, οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις σε κεφάλαιο, αλλά επενδύουν και σε εργαζομένους και σε ανθρωπίνους πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη ασφάλεια για τις επιχειρήσεις μας μεν, αλλά πρέπει να γίνει και ένας κατάλληλος συσχετισμός ε, και με το κοινωνικό μοντέλο και να το συνδυάσουμε και αυτό με τις συμβάσεις εργασίας, γιατί έτσι θα ευνοηθούν πολλοί παράγοντες. Επίσης, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, γιατί αναφερθήκατε ακροθυγός αυτός, ε, στην έλλειψη των επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς ε, προκειμένου να δώσουμε κίνητρα, ώστε οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επανέλθουν στα προσδοκάμενα επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας έχει ξεπεράσει, για παράδειγμα, η Κίνα ε, πάρα πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν επενδύουν πια ε, παρά μόνο ένα 2% του κύκλου εργασιών τους σε έρευνα και ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Ωραία. Τέσσερα λεπτά για τους κυρίους και τεσσεράμιση λεπτά για τις κυρίες. Αυτό προτείνατε, δεν είναι. Από το ECR, ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπιανκόφσκα, ορίσατε στη συνεδρίασή μας και σας ευχαριστώ για τη σημερινή σα παρουσία εδώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το τμήμα σας ε, για την βοήθεια που προσφέρει στις μικρές επιχειρήσεις στην περιφέρειά μου. Σπανίω ε, ε, ευχαριστούν επιτρόπους οι Βρετανοί συντηρητικοί, αλλά να ορίστε που συνέβη και αυτό. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τελωνιακό κώδικα και εγώ συναντήθηκα με τον κύριο ε, Καλέα, ο οποίος είναι στην αίθουσα εδώ σήμερα και χάρη σε αυτές τις συναντήσεις το πρόβλημα επιλύθηκε. Για ε, μία φορά λοιπόν βοηθήσατε μια μικρή επιχείρηση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα να περάσω στην παρουσίασή σας. αναφερθήκατε διαμακρών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευπρόσδεκτο αυτό μεν, αλλά διαπίστωσα ότι έχουμε πολλά ωραία λόγια και ελάχιστες συγκεκριμένε προτάσεις. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να σας προτείνω είναι η βιομηχανία, είτε είναι μικρή είτε μεγάλη, δεν χρειάζεται μεγαλό σχέδιο από την Ευρώπη. Χρειάζεται να τις επιτρέψουμε να απασχολεί ανθρώπους, να δημιουργεί θέσει εργασίας και ευημερία και ανάπτυξη εκ του μηδενός. Και πραγματικά φρονώ ότι το πρόβλημα είναι η υπερβολική Ευρώπη και όχι η λίγη Ευρώπη και το τμήμα σας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη, θα μπορούσε να μας κάνει μια τη χάρη να ανακαλέσει την νομοθεσία και να μην επανέλθει με, κιά, με άλλες περίπλοκες προτάσεις. Πραγματικά λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και ε, σας έθεσα την ίδια ερώτηση και στην ακρόασή σας ε, για να αναλάβετε καθήκοντα πριν από μερικούς μήνες. Σας ρώτησα ποιο νόμο ε, ευρωπαϊκό κατά πάσα πιθανότητα θα ανακαλέσετε και δεν μπορούσα να θυμηθείτε το έναν. Κυρία Επίτροπε, τώρα είστε Επίτροπος για περίπου ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο, λέει ο μιλητής. Ελπίζω λοιπόν ότι αφού διατελέσετε επίτροπος για κάποιο διάστημα θα έχετε σκεφτεί κάποιο νόμο το οποίο θα μπορούσαμε να διαγράψουμε. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι αυτός. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Δεμπάκερ, εξ ονόμους του Στουάλτε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και από πλευρά μα κάποιε ερωτήσει. Να ευχαριστήσουμε καταρχά την Επίτροπο για την επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή μα. Και να πω και ότι και εγώ από πλευρά μου και το λέω πάντα στιευόμενος αυτό, ότι η γενική σας διεύθυνση είναι αυτή που γράφει τις καλύτερες λευκές, πράσινες βίβλους, τις καλύτερες επιστολές, αλλά τελικώς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή. Και ακριβώς αυτό είναι και ο στόχος της ερώτησής μου. Ξέρετε ότι για πολλές από τις πρωτοβουλίες που αναφέρετε στην επιστολή σας χρειάζεται τουλάχιστον μια χείρα βοηθείας, αν όχι και το μεγαλύτερο έλεγχο από πλευράς κρατών μελών. Και θα ήθελα να ξέρω τι μόχλευση πιστεύετε ότι έχετε ενώπιον των κρατών μελών και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να, να συνεργαστείτε μαζί τους καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, ώστε πραγματικά να καταλήξουμε σε κατάλληλη νομοθεσία. Ο κύριος Φόξ είπε ότι ίσως χρειαζόμαστε λιγότερο Ευρώπη. Ε, όποια νομοθεσία γίνεται εδώ ε, εγκρίνεται τουλάχιστον από τα κράτη-μέλη και από το δικό σας κράτο μελους Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε καλύτερη νομοθεσία, πού μπορούμε να έχουμε πραγματική προστιθέμενη αξία της Ευρώπης και πώς μπορούμε να πείσουμε ε, τα κράτη-μέλη για την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Ε, πώς σκοπεύετε λοιπόν να ε, έχετε και τα κράτη-μέλη με το μέρος σας. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και επίσης ένα τμήμα της πολιτικής σας είναι η ενεργειακή πολιτική. Ξέρω ότι δεν είναι 100% δική σας αρμοδιότητα, αλλά επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία στο διεθνές προσκήνιο. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση για την ενέργεια. Ποια είναι η άποψή σας, τι λείπει από βιομηχανική σκοπιά και δεύτερον, εμείς, ή μάλλον η Επιτροπή, προετοιμάζει μια νέα πρόταση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, και θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση βεβαίω και στην Επιτροπή μα. Ε, θα ήθελα και κάποιε απόψει από εσά, γιατί δεν αναφέρετε τίποτα στην επιστολή σα. Ποια είναι η πρώτη σα άποψη, τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα, ώστε να αντισταθμίσουμε το γεγονό ότι έχουμε, θέλουμε να έχουμε μια πιο πράσινη οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Και επίση, διαπιστώνουμε ότι πολλέ επιχειρήσει που έκαναν επενδύσει τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιούν τεχνολογία εχμή και μπορούν να γίνουν καλύτεροι με τις ε, ε, ε, εξελίξεις της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ώστε να ανταμυφθούν κατά κάποιο τρόπο με το νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών, ώστε να μην χρειαστεί να αγοράσουν τα αρχικά δικαιώματα εκπομπών και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς και ίσως και καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την κείμενη νομοθεσία γίνονται πολλές αλλαγές στην οικονομία μας. Περνάμε από μια οικονομία που βασίζεται σε προϊόντα σε μια οικονομία που βασίζεται κυρίως σε υπηρεσίες. Και αυτό φυσικά έχει και επίδραση στην ε, βιομηχανία. Ε, αλλάζει νοοτροπία, ασχολούμαστε με τις υπηρεσίες, αντανακλάται και στην κυκλική οικονομία, αλλά αυτή τη στιγμή παρακολύεται και από πολλές εθνικές νομοθεσίες αλλά και από την ίδια την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχετε κάποιο άποψη για το τι θα μπορούσε να δουν, ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες, διότι υπάρχει αυτή η μετατόπιση και θα ήθελα... Ε, νομίζω να γνωρίζουν και οι πολίτες μας ε, πώς ε, γίνεται οι μικρές επιχειρήσεις, πολλές φορές νεοφυείς επιχειρήσεις να βρουν ένα περιθώριο ε, για να δραστηριοποιηθούν και αυτές και να φροντίζουμε να παρέχονται συγκεκριμένε υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτά από μένα και περιμένω συγκεκριμένε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Μπουτικόφερ, εκ μέρους των Πρασίνων, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε σε πολλά με τα οποία συμφωνώ και πιστεύω πως συμφωνούμε όλοι. Για παράδειγμα, το ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός ε, στην ε, καινοτομία και σε άλλους ε, τομείς των βιομηχανικών εξελίξεων. Επίσης, κατανοούμε ότι δεν πρέπει να επιλέξουμε μια στρατηγική που θα κλείσει πόρτες, αλλά που θα ανεβάσει τον πύχη ε, σε σχέση με την αλυσίδα αξιών, με την προώθηση της καινοτομίας, με την... Ε, με το να αρθούν τα διάφορα εμπόδια και όλα αυτά περιέχονται στην ανακοίνωση του 2011 και ε, ορθώς αναφέρονται αυτά. Ελπίζω να συνεχίσετε να επιδιώκετε τους ε, στόχους αυτούς. Αυτό όμως που δεν άκουσα και δεν βλέπω είναι πολιτικές οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Αυτό που δεν βρήκα πουθενά, που δεν άκουσα πουθενά, είναι κάποιες ε, συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό πρόβλημα που έχουμε. Δεν έχουμε ευρωπαϊκή ε, πολιτική, βιομηχανική πολιτική, διότι δεν υπάρχει η αρμόδια ευρωπαϊκή ε, πολιτική αρχή. Πώς λοιπόν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη για να δημιουργήσουν σύγχρονη καινοτόμο τεχνολογία στην βιομηχανία όταν τα κράτη-μέλη δεν ε, έχουν κάποιον ε, φορέα που να τους εκπροσωπεί. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν την Ευρώπη προς το καλύτερο αλλάζοντας αυτό ακριβώς ε, το, αυτή, αυτήν ακριβώς την έλλειψη. Και ελπίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Φόξ ότι δεν θα παραμείνουμε μόνο σε αυτά τα καθιστικαστικά λόγια αλλά θα έχουμε και πράξεις και τώρα, αυτά ήταν ε, τα πράγματα με τα οποία συμφωνούσα. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία με βρίσκουν αντίθετο. Μιλήσατε για την ανταγωνιστικότητα. Αλλά αυτό που δεν αναφέρατε καθόλου είναι το ότι αυτή εδώ η Επιτροπή πέρυσι, ή μάλλον όλο το Κοινοβούλιο πέρυσι, συμφώνησε να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία θα συνδυάσει την βιωσιμότητα με την ανταγωνιστικότητα και στην παρουσίασή σας μας είπατε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίφαση με την βιομηχανική πρόοδο και με, την, με το κλίμα, αλλά μόνο όταν συνδυαστούν αυτά θα έχουμε μια επιτυχημένη βιομηχανική ε, πολιτική. Και επίσης σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και δεν άκουσα να αναφέρετε ούτε τα συνδικάτα ούτε τους ε, εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί πιστεύω πως ε, και εκείνοι έχουν να συνεισφέρουν και πρέπει να συνεισφέρουν, διότι όταν θέλουμε καινοτομία, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι μεν ένα από τα πιο δυνατά μέσα που έχουμε, αλλά η καινοτομία δεν ε, πραγματοποιείται από κανέναν άλλον παρά από το εργατικό δυναμικό. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε φωνή και βήμα σε αυτό το εργατικό δυναμικό και αυτό δεν το άκουσα στην παρουσίασή σας. Επίσης, σήμερα το πρωί παραβέθησα σε ένα συνέδριο για, την, ε, για τον κατασκευαστικό τομέα και δεν αναφέρθηκαν ε, ποτέ, δεν αναφέρθηκε ποτέ η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ε, νομοθετικού πλαισίου που θα δώσει ε, όθηση και πρόθεση στην βιομηχανία. Πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι ως προς ε, την πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Βλέπω ότι υπάρχει μια καινούργια προσέγγιση, μια καινούργια φιλοσοφία. Δεν την ε, βλέπω όμως με τα μάτια μου. Και ελπίζω αυτό να μην είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Σιλικιώτης τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς με τη σειρά μας να καλωσορίσουμε την κυρία Μπιεσκόφσκα εδώ στην Επιτροπή μας. Βεβαίω ακούσαμε πάρα πολλά. Κατά την άποψή μας, εάν δεν δούμε πραγματικά τις αιτίε της κρίσης και της αποβιμηχανοποίησης που δεν είναι άλλες από τις πολιτικές της αυστηρής λιτότητας οι οποίες προωθήθηκαν και συνεχίζουν να προωθούνται σε πολλά κράτη-μέλη, οι οποίες ουσιαστικά είναι πολιτικές που λειτουργούν ηφαισιακά και αντιαναψυκτιακά διότι είναι οι πολιτικές που διέλυσαν τον βιομηχανικό τομέα ιδιαίτερα στον Νότο. Ζούμε στον Νότο της Ευρώπης μια ε, σχεδόν ε, μεγάλη αποβιομηχανοποίηση, μειώθηκαν επενδύσεις, ταυτόχρονα παραβιάζονται θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, οδηγούν στο κλείσιμο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταδικάζουν στην αργία εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι να προωθήσουμε μια ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική χωρί αποκλεισμού, που απότερο στόχο πρέπει να είναι να αντιμετωπίσει την ανεργία, ιδιαίτερα ανάμεσα στου νέου, να δημιουργήσει νέε ποιοτικέ θέσει εργασία, οι οποίε βεβαίω να είναι ασφαλεί και αξιοπρεπεί ε, και να οδηγήσει σε μια βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη. Κατά τη δική μα άποψη, η, η ανάπτυξη αυτής της ατζέντας για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, θα έχει αξία μόνο να γνωρίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, οι πολιτικές που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των προβλημάτων, που δεν είναι άλλες από τις νεοφιλεύθερες πολιτικές και να στηριχτεί πάνω σε νέους άξονες. Πρώτον, για μας χρειάζεται να υπάρχει αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και το κράτος ο, ο, τα κράτη οφείλουν να στηριχτούν από την Ευρωπαϊκή για να οδηγήσουν σε δημόσιες επενδύσεις και το δεύτερο είναι να επανεξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα θεσμικά όργανα την πολιτική των κρατικών επιδοτήσεων. Είναι ένα ζήτημα που φέρνει σε μειονεκτική θέση την ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στη βιομηχανία άλλων χωρών και περιφερειών. Και επειδή θέτουν το ερώτημα, το ζήτημα που είπαν και μερικοί προηγούμενοι συνάδελφοι από το ΙΣΙΑ και την Άρτε, το θέμα δεν είναι περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους είναι ποια Ευρώπη θέλουμε. Ε, και εμείς θέλουμε μια Ευρώπη ε, περισσότερο κοινωνική, αναπτυξιακή ε, που να διασφαλίζει πρώτα απ' όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων και τις αξίες των ίδιων των ανθρώπων. Και εδώ κυρία Πιεσκόφσκα δεν κατάλαβα αυτό που θέσατε ως παράδειγμα για την βιομηχανία με τις 500 θέσεις μηχανικών με υψηλά προσόντα και ερευνητών δεν κατάλαβα ποιο ήταν το νόημα. Δηλαδή θα προωθήσουμε την αντίληψη, διότι αυτή είναι η αντίληψη που δημιουργά περαιτέρω προβλήματα, να ενισχύσουμε την αντιγωνιστικότητα διαλύοντας τις εργασικές σχέσεις, περιορίζοντας ε, τα εργασιακά δικαιώματα ε, και τους μισούς ακριβώς είναι αυτό που δεν θέλουμε ακριβώς γιατί μια τέτοια ε, βιομηχανία θα στηρίζεται σε λαθασμένες βάσεις σε ξύλινα ποδάρια και όχι σε στέρεες βάσεις σωστών εργασιακών ε, σχέδιων που θα στηρίζονται στις συλλογικές συμβάσεις που θα ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το επόμενο, ενώ βλέπουμε να, να προωθούνται συνεχώς μέτρα σε χώρε που υπάρχει κρίση για ενίσχυση του τραπεζικού, του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν βλέπουμε μέτρα. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αυτό. Ποια μέτρα θα ε, πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει ε, τη βιομηχανία, ιδιαίτερα στις χώρες που μαστίζονται από την κρίση. Μιλήσατε κυρία Επίτροπε για την έρευνα και την καινοτομία. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε να μειώνονται τα κονδύλια στο budget ε, για την έρευνα και την τεχνολογία. Ε, επίσης το ερώτημα και τελευταίο αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα ποια μέτρα θα πάρουμε ώστε οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν το των ανταγωνισμών εφόσον περάσει η συμφωνία ε, για διατλαντικές επενδύσεις και εταιρική συμφωνία γνωστή TTIP οι θα ακυρώ, αυτή η συμφωνία θα αφαιρέσει κανονιστικές διατάξεις και θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, thank ευχαριστώ πολύ κύριε Συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπορέλη, εκ μέρους της ομάδας EFTD. Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την επιστολή σας, ε, ιδιαίτερα το παράρτημα. Στην τρίτη ενότητα του παραρτήματος, με τίτλο «A Business Friendly Environment», γίνεται μνήα σε μια σειρά από παρεμβάσεις, ε, περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκες, για να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε πίστοση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ ωραία. Πριν όμω αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, τα οποία μπορεί να είναι και πολύ καλά διαρθρωμένα, γιατί να μην μιλήσουμε για την αποτελεσματική εφαρμογή ενό ε, μέσου ευρωπαϊκού, το οποίο είναι πολύ καλά θεσπισμένο, ε, για την καθυστέρηση πληρωμών. Ε, ένα μέσο το οποίο, άμα τεθεί σε αποτελεσματική εφαρμογή, θα δώσει μια ανάσα ζωή στι μικρομεσαίες επιχειρήσει και θα βοηθήσει και την, ε, τις πιστώσεις. Μέχρι το Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να υποβληθεί μια έκθεση για την εφαρμογή αυτή τη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να ε, υπάρχουν και μια σειρά από ε, βέλτιστες προτάσει. Τι μπορείτε να μα πείτε λοιπόν για την παρακολούθηση αυτή τη οδηγία και τι ιδέε που πρέπει να παρουσιαστούν. Επειδή η οδηγία ε, από το 2013 επιβάλλει μια καθυστέρηση το μέγιστο 30 ημερών για την υστέρηση πληρωμών και σε πολλές μέρες, όχι μόνο στην Ιταλία, σε πολλές χώρες είναι πάνω από 160 ημέρες αυτή η καθυστέρηση. Αυτά είναι στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη σχετική Γενική Διεύθυνση. Και σε όλε τι περιπτώσει των καθυστερήσεων, οι καθυστερήσει είναι από τη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν επιχειρήσει στην Ιταλία, το 60% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι δεν υπήρξαν θετικέ συνέπειε από τη συγκεκριμένη οδηγία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πλήττει την ίδια την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άποψη έχετε εσεί. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά την το νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα Φαίνεται ότι αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τι επιχειρήσει που θέλουν να καταχωρήσουν το, την εφεύρεσή του και για τι 28 χώρε μέλη. Επειδή υπάρχει μεγάλο κόστο όμω ε, διατήρηση αυτού του διπλώματο ευρεσιτεχνείου, τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη που προτιμούν να υπάρχει μια πιο περιορισμένη εφαρμογή. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ έχει το λόγο πρώτη φορά στην ιστορία της Επιτροπής μας για την νέα ομάδα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε για την παρουσίασή σας. Δείξατε μια ισχυρή δέσμευση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και για την ανταγωνιστικότητα αυτής. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα με τους τρεις κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δηλαδή μια ενσωμάτωση της, της ε, ε, αξιών, φιλική προς το περιβάλλον και με έμφαση στην καινοτομία. Σίγουρα είναι ένα πολύ καλό όραμα για την Ευρώπη και γι' αυτό το στηρίζουμε. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο για το μέλλον και εύχομαι να το καταφέρετε. Έπειτα αναφερθήκατε και στην συνεκτίμηση της ε, διάστασης ε, της ε, βιομηχανίας στην κοινοτική πολιτική της, Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και κάτι που μάλιστα η Ιταλική Προεδρία προσπάθησε να δρομολογήσει. Αναφερθήκατε επίσης και στη σημασία της ψηφιοποίησης, η οποία σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να αναπτυχθεί πολύ ε, γρήγορα η βιομηχανία. I think it works now. Νομίζω πως λειτουργεί το σύστημα τώρα. Παρακαλώ, αρχίστε από την αρχή. Λοιπόν, δώσατε λοιπόν μια συνέντευξη στη Handelsblatt όπου αναφερθήκατε στην μεγάλη σημασία της ψηφιοποίησης, αναφερθήκατε κατά της υπερβολικής νομοθεσίας και είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε ελευθερία στις επιχειρήσεις. Επίσης τονίσατε τη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης και πώς πρέπει να ενσωματωθούν όλα αυτά στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αναφερθήκατε επίσης στην στρατηγική Ευρώπη 2020 και στο ότι η παραγωγή πρέπει να παραμείνει ε, στα... στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα πολλές φορές είναι τελείως διαφορετική. Τα τελευταία πέντε χρόνια χάθηκαν 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Μειώθηκε κατά 6% η απασχόληση. Μειώθηκαν οι άμεσες επενδύσεις. Η διπλασιάστηκε η φορολογία. Είναι τώρα διπλάσια από τη φορολογία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυξήθηκαν οι τιμές ε, των, ε, της ε, ενέργειας. Και πάλι κατά το διπλάσιο υψηλότερες από τις στις Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη είναι στην τέταρτη θέση ε, την καινοτομία. Και μας αναφέρατε την ανάγκη για αύξηση της ψηφιοποίησης. Όμως εγώ βλέπω πάρα πολλά κενά στις προτάσεις σας. Όλο ένα και αποδυναμώνεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία και όλα αυτά σε συνδυασμό έχουν οδηγήσει σε μια ανάγκη 400 ε, δισεκατομμυρίων ε, ευρώ στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που εσείς προτίθεστε να εφαρμόσετε έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο παγκόσμιο στερέωμα, ιδιαίτερα έχοντας ως αντίπαλο την ε, Κίνα ή και την ε, Ιαπωνία ακόμα. Ποια μέτρα σκοπεύετε να εφαρμόσετε και πώς θα δώσετε κίνητρα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να συνεισφέρουν με την ε, σειρά τους τη δημιουργία ενός ικανού πλαισίου που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνετε με τη φορολογία, τι θα κάνετε με τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και τι θα κάνετε με τις ε, διαδικασίες ε, αδειών για την ε, ενέργεια. Τι θα κάνετε λοιπόν για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και ποια μέτρα θα, αναλάβει η Ευρωπαϊκή, θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ. Ήταν πολύ μακρά αυτή η παρέμβαση. Διακόπιν πολύ. Λοιπόν, εντάξει, συνεχίσατε. Καλώς δεν υπάρχει, δεν έγινε και τίποτα. Αν επιτρέπετε, συνάδελφοι, να προτείνω στην Επίτροπο την κυρία Πιανκόφσκα να απαντήσει, διότι τουλάχιστον είχε τρεις με τέσσερι ερωτήσεις από κάθε ομιλητή. Οπότε είναι πολλές ερωτήσεις Καλό να αρχίσει να απαντά και μετά θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος ερωτήσεων και σχολείων. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. κάποια από εσά. Τέλο πάντων, θα προσπαθήσω να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Αν κάποιε ερωτήσει όμω έχουν επαναληφθεί, θα προσπαθήσω να καλύψω μαζί. Πρώτα απ' όλα, κάποια αξιότιμα μέλη έθεσαν το εξή ερώτημα. Ποια συγκεκριμένα μέτρα επί ποιων συγκεκριμένων θεμάτων θα κινηθούμε και θα εργαστούμε. Καταρχάς επαναλαμβάνω. Θέλω τις λιγότερες δυνατές νομοθετικές προτάσεις. Εμείς στην υπηρεσία μου έχουμε αποσύρει τις περισσότερες προτάσεις. Προσπαθήσαμε να βρούμε ποια είναι τα καλύτερα θέματα να επεξεργαστούμε στους επόμενους μήνες. Θα επεξεργαστούμε ό,τι έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυτό που είναι επιζήμιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ο κατακαιρματισμός. Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, προδιαγραφές, αμοιβέ αναγνωρίσεις, πλατφόρμες, πρότυπα και επιβολή των νομοθεσιών. Πολύ ισχυρή προσπάθεια σε αυτό. Επαναλαμβάνω αυτό που ήδη έχω πει. Πολύ σωστή υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι σημαντικότατη κατά την άποψή μου. Τα πρότυπα και προδιογραφές σημαντικότατα και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Για το διάστημα πρέπει να εστιαστούμε επί δύο προτεραιοτήτων. Έχουν το, στο Γαλιλαίο και στο Κοπέρνικος. Έχουν μεγάλη προτεραιότητα. Εκτοξεύθηκε το Sentinel 2α του Κοπέρνικος μαμε δορυφόρο δορυφόρος 2α, πηγαίνουμε πολύ καλά. Ο Γαλιλαίο το 2016 θα αρχίσει να δίνει πρώτες υπηρεσίες, θα είναι πλήρω λειτουργικό το 2020. Αυτά είναι πολιτικά προγράμματα. Εστιάζονται σε πολιτικέ υπηρεσίε όσον αφορά το Γαλιλαίο. Όμω, είναι σημαντικό ο Γαλιλαίο και για την άμυνά μα. Η κυρία Νίμπλερ έθεσε ένα άλλο ερώτημα για τις ε, ε, επαφές μας και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ήταν και καλύτερες και χειρότερες οι σχέσεις με την πάδο των ετών. Εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος όπως και άλλα κράτη-μέλη και άλλες χώρες. Όμως πληρώνουμε σημαντικά ποσά Οπότε πρέπει να έχουμε πραγματικά καλή επαφή με τον φορέα αυτό και θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά που θέλουμε να κάνουν. Υπάρχει έλλειψη επενδύσεων. Και γι' αυτό απευθύνω έκκληση και σε εσά, διότι για την ΕΦΣΗ, στο ΕΦΣΗ, στο πρόγραμμα στατικές επενδύσεις, έχουμε μόνο μερικές χιλιάδες προγράμματα που παρέχονται από τα κράτη-μέλη. Ε, δέκα από αυτά αφορούν τη βιομηχανία μόνο. Και θα ήθελα να έχω δρομολογηθέντα βιομηχανικά τέτοια προγράμματα και σχέδια, όχι μόνο υποδομές. Πριν πρόσφατα είχαμε ένα πρόγραμμα που είχαν υποβάλει και όλα τα κράτη-μέλη, τώρα έχουμε δέκα. Αλλά είναι ακόμα πολύ μικρός αριθμός εν συγκρίση με τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εδώ έγκυται και ο δικός σας ρόλος, κατά κάποιο τρόπο. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έρχομαι σε επαφές με τα κράτη-μέλη και δεν λειτουργούν τέλεια τα πράγματα εκεί και θα προσπαθήσω μαζί με τις προεδρίες, με την Προεδρία του Λουξεμβούργου που θα αναλάβει να έχουμε πολύ καλύτερη συνεργασία στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, άρα και καλύτερα αποτελέσματα. Και θα πω μερικά λόγια και για τα βιομηχανικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΥ, διότι εδώ είναι η ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Προγράμματα για την ενεργειακή απόδοση, Φερρυπίν. Μου έρχεται έτσι στο μυαλό όταν σκέφτομαι βιομηχανικά προγράμματα αυτό. Αλλά υπάρχει μεγάλη έλλειψη προτάσεων από τα κράτη-μέλη. ετέθησαν κάποιες ερωτήσεις για το παράδειγμα που σας έδωσα. Να σας πω ότι αναφερόμουν σε αυτό που μου είπαν λίγες εταιρείε για την ευελιξία. Εγώ νοιάζομαι για κοινωνικά θέματα και πολύ. Το συζητήσαμε στο κολέγιο της Κομισιόν, αλλά θέλω να ακούσω και τι λέει η βιομηχανία και τι λένε οι εταιρείε. Τι μας λέει η βιομηχανία, μας λέει ότι υπάρχει έλλειψη ευελιξίας στην Ευρώπη. Εάν θέλουμε, αν υπάρχει ευκαιρία να κερδίσουμε λίγες θέσεις εργασία που απαιτούν πολύ ψηλά προσόντα για 2, 3, 5 χρόνια, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι καλύτερο να τις έχουμε αυτές στην Ευρώπη. Βέβαια με όλα τα συναφή εργασιακά δικαιώματα παρά όμως να μην, έχουμε, να μην έχουμε εμείς εργασίες και να φύγουν και να πάνε Κίνα και Αμερική, καλύτερα να τις έχουμε εμείς. Και το θέματα των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της παιδείας, αυτό το επαναλαμβάνουν συνεχώς επιχειρήσεις, ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και δεν ταιριάζει το επίπεδο της παιδείας, η παιδεία που παρέχεται, που παράγεται από τα πανεπιστήμια και των αναγκών της βιομηχανίας, των δεξιοτήτων, ικανοτήτων γνώσεων που ζητάει η βιομηχανία έρευνα και ανάπτυξη. Εκεί ετέθησαν ερωτήσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλά χρήματα σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτά τα χρήματα όμως, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αφορά τις εταιρείες που αποκαλούνται παραδοσιακές, ούτως υπήν. Υπάρχει, υπάρχει πλήρης έλλειψης ανάληψης κινδύνου από τις τράπεζες. Δεν θέλουν να χρηματοδοτούν τις καινοτόμες εταιρείες. Οι καινοτόμε εταιρείε πρέπει να ψάξουν να βρουν χρήματα εκτό Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα από του στόχου μα, να το αλλάξουμε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που θα παρουσιαστούν στην Ένωση των Κεφαλαγορών. Εμείς δεν είμαστε πιο ανόητοι από άλλα μέρη στον κόσμο. Γιατί να μην δημιουργήσουμε εταιρείε που είναι πραγματικά καινοτόμε, που να μπορούν να αναπτύσσουν να αναπτυχθούν από 0 μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε 2 εκατομμύρια ανώτατο όριο στην Ευρώπη. Μέχρι εκεί μπορούν να πάρουν χρήματα οι εταιρείε. Για παραπάνω πρέπει να στραφούν στο εξωτερικό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Συμφωνώ με τον κύριο Φόξ. Συμφωνώ. Θέσει εργασία δημιουργούνται από εταιρείε και όχι από τη δίκηση και τι κυβερνήσει. Συμφωνώ με αυτά που είπατε λιγότερες ρυθμίσεις, λιγότερη νομοθεσία, λιγότερο βάρος στις εταιρείε, λιγότερη φραγμή. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, πρέπει να ακούσουμε τη λέει βιομηχανία. Και θέλω να πω ξανά ότι εμείς και οι υπηρεσίε μου αποσύραμε τα περισσότερα νομοθετήματα όταν έγινε αυτή η προσπάθεια τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο φέτος. Συμφωνώ επίσης και εμένα δεν μου αρέσουν τα μεγάλα σχέδια. Λοιπόν, 8 μήνες είμαι σε αυτή τη θέση, όχι σχεδόν ένα χρόνο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες σκέψεις επί χάρτου. Αλλά παρακαλώ κρίνετε εμέ και τις ε, υπηρεσίες μου από αυτά που θα πετύχουμε, από το έργο μας. Τι βλέπω σαν βασικό και απευθύνομαι σε κάποιους από εσά, για τη βιομηχανία κυρίως, για τη μεγάλη βιομηχανία που έχουν ε, επενδυτικά σχέδια μακρά πνοή. Θέλουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα τη νομοθεσία οι μεγάλε επιχειρήσει. Αυτό ζητούν. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν να πετυχαίνουν επίπεδο για κάτι που θέλουν να παράξουν και εμεί να θεσπίσουμε νέα νομοθεσία σε αυτή τη φάση που κάνει, απομακρύνει το στόχο χρονικά. Και αλλαίως πώς. Επίσης, πρέπει να πω και δύο λόγια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκύπτουν και από την εθνική νομοθεσία, φορολογία, ίδρυση εταιρεία ε, και επίσης σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα νομοθετήματα που έχουμε σε εθνικό επίπεδο και όχι τα ευρωπαϊκά. Ε, θα προσπαθήσουμε όμως να τα δούμε ανακλάδο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε σε αυτό, αλλά ο πρώτος κλάδος θα είναι σίγουρα ο κλάδος της χημίας, διότι έχει πληγή από την πολύ αναλυτική ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σίγουρα να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Μπουτικόφερ, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη να τα δούμε τα πράγματα από την αρχή. Δεν ε, αναφέρθηκα απλώς στη βιωσιμότητα. Είπα ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα. Νομίζω ότι αυτό ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε σίγουρα ε, μιλάμε με όλους τους ενδιαφερομένους, εξετάζουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο. Ε, υπήρχε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τις ενεργοβόρες ε, βιομηχανίες και εκεί είχαμε εκπροσώπους της βιομηχανίας, ε, περιβαλλοντικών με κυβερνητικών οργανώσεων και των συνδικάτων. Δεν μιλάω μόνο με τη βιομηχανία, αλλά μιλάω με ε, μια ευρία ομάδα ανθρώπων που έχουν πολλά πράγματα να πούνε για την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την βιομηχανική βιωσιμότητα θα συνεργαστώ στενά με τα κράτη-μέλη στα θέματα της εφαρμογής και στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα και ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, σίγουρα δεν είναι τέλεια Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αλλά και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών. Διότι όπως ε, βλέπω εγώ τα πράγματα τώρα, με αυτή τη φρέσκια ματιά που έχω, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία δυστυχώς σε επίπεδο Συμβουλίου. Για τις πολιτικές, για τις κρατικές ενισχύσεις θα σας απαντήσω γραπτός. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι κρατικές ενισχύσεις ε, και η ενέργεια είναι ε, δύο θέματα τα οποία συζητούν και ο Επίτροπος Κανιέτε και ε, ο άλλος αρμόδιος Επίτροπος. Πρόκειται για τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη βιομηχανική πολιτική και σίγουρα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας και ήδη συνεργαζόμαστε. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δείχνει τη δική μας προοπτική και προτείνει κάποιες λύσεις για τις κρατικές ενισχύσεις από τη βιομηχανική σκοπιά και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τα δούμε τα πράγματα και από αυτό το πρίσμα, όπως και οπουδήποτε αλλού. Αν μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει κάτι αυτό το οκτάμινο, έχουμε καταφέρει να ε, εξορθολογήσουμε τα θέματα της βιομηχανίας και να περάσει σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρει και η άποψη της βιομηχανίας σε όλες τις στρατηγικές και σε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά. On, on financial για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Είπα δυο λόγια να πω κάτι ακόμα ε, για το ενίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ε, διότι υπήρξε και μια ερώτηση από αυτού. Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόλις συζητήθηκε σήμερα στην, ε, επιτροπή, στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών υπήρχε μια αρκετά κρέα στάση από κάποια κράτη-μέλη να είναι πολύ υψηλά τα τέλη ανανέωση του διπλώματο ευρεσιτεχνία. Δηλαδή αυτά τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται ετησίω ε, για την ανανέωση του διπλώματο ευρεσιτεχνία. Απέστειλε επιστολή σε όλου του υπουργού. Ε, με κάποιους συνομίλησα και τηλεφωνικούς εχθέ, ε, διότι ορισμένε φορέ ε, υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη που είναι υπέρ της ενίας αγοράς και της ελεύθερης αγοράς και ε, μου ζήτησαν να έχουμε πολύ υψηλά τέλη ανανέωσης. Ε, δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη λύση σήμερα, αλλά ο λόγος για τον οποίο υπήρξε όλη αυτή η διαμάχη είναι γιατί τα τέλη ανανέωσης εν μέρη είναι κόστος το οποίο επιμερίζεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνών και το Εθνικό Γραφείο Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και τα Εθνικά Γραφεία ζητούσαν πολύ ψηλά ετήσια τέλη. Δεν ξέρω τι απόφαση λήφθη σήμερα, αλλά επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω και γραπτός. Εάν ε, ε δεν καταφέρουμε να έχουμε χαμηλά τέλη ανανέωσης, ε, με πολύ χαμηλά τέλη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί εγώ αυτό είχα προτείνει. Σας ευχαριστώ. Uh, oh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Παίρνουμε τώρα στον ε, δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, τα μέλη της Επιτροπής μας. Θέλω να σας προτείνω κάτι. Να μην μιλήσετε παραπάνω από δύο λεπτά, γιατί έχω δέκα ονόματα στον κατάλογο των ε, ομιλητών και πρέπει να τελειώσουμε στις πέντε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιοριστούμε στα δύο λεπτά. Πρώτος ο η κυρία Κόμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Επίτροπο για τη σημερινή της παρουσία εδώ, γιατί αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ χρήσιμες για μας. Θα κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά το ε, με την, ε, στο οποίο είστε πολύ δραστήρια. Όσον αφορά το άρθρο 5 της πρότασης κανονισμού, άρθρο 7 συγγνώμη, εγώ είμαι και συγγήτρια για την εποπτεία της αγοράς και θα ήθελα να μου πείτε δύο ε, πολύ γρήγορα πράγματα. Καταρχάς, αν μπορείτε να συμπεριλάβετε, επειδή αυτοί οι δύο τομείς ο τομέας των κοσμημάτων και της επίπλωσης που είχαν δώσει θετικές νομοδοτήσεις και ήθελαν να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κανονισμό με την και αν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε το πράσινο φως και το δεύτερο σχετίζεται με τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο εξακολουθεί να αντιτίθεται στο θέμα του made in, ε, του κατασκευασμένου στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε μια εκτίμηση αξιολόγηση επιπτώσεων. Πάρα πολλές χώρες και η κλάδοι είναι υπέρ αυτών των προϊόντων προέλευση και για, τις, για προϊόντα εκτός των τροφίμων και θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν δίνονται ε, λοιπόν το πράσινο φως για αυτή την περίπτωση. Ένα λεπτό μίλησα, οπότε έχει χρόνο ε, ο επόμενος ομιλητής να μιλήσει περισσότερο. Okay, sorry. Μάλιστα, άκουγα ακόμα τη διερμηνία. Επόμενος ομιλητής, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπη, η... η νέα εκβιομηχάνηση έχει σκοπό να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγαθών στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό, όμως υπάρχει επίσης και το outsourcing. Και μάλιστα στον τομέα αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές ε, καινοτόμες ε, ιδέες και προτάσεις Και αυτή ίσως είναι μία απάντηση σε όσους προκάλεσαν την απόβιο ε, απόβιομηχάνηση. Υπάρχουν πολλές ε, νέες καινοτόμες ευρεσιτεχνίες, πολλά νέα εργαστήρια, μέθοδοι κατασκευής κτλ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς θα στηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν υπάρχουν αυτοί οι δισταγμοί από πλευρά κρατών μέλων. Πώς θα εφαρμόσετε λοιπόν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο στην περίπτωση που το κεφάλαιο είναι αυτό που αποφασίζει τι θα γίνει με τις ε, τοπικές επενδύσεις. Γιατί μας είπατε ότι όλα πρέπει να είναι δικτυωμένα και να συμβαίνουν και να αλληλοσυνδέονται, όμως εγώ δεν το βλέπω αυτό. Μας είπατε επίσης ότι δεν μπορεί ένα και μόνο εργοστάσιο να πραγματοποιήσει όλα τα στάδια της παραγωγής. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Πολμπάτσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία πίτροπε για το ότι ήρθατε εδώ και μας κάνατε αυτήν την ε, παρουσίαση για την ε, ολιστική προσέγγιση του θέματος της βιομηχανίας. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στις ε, καινοτομίες. Έχω στα χέρια μου ε, την νεότερη μελέτη για τις ε, καινοτομίες και βλέπω ότι το κόστος της καινοτομίας είναι πολύ ψηλό και αποτελεί εμπόδιο Είναι λοιπόν εμπόδιο το κόστος τη καινοτομία ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά νέε καινοτομέ μεθόδους. Υπάρχουν επίσης αυτά τα ποσοστά που βλέπω για, που έχουν σχέση με τις ελλείψει. και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχουμε τον ορίζοντα 2020, έχουμε τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που σκοπό έχουν να ενισχύσουν και να τονώσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από αυτά για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόστου, του διοικητικού φόρτου, της εγγραφειοκρατία. Τι προτίθεται λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελαφρύνει το φορτίο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τις γλιτώσει από την καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέρνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ την κυρία Βιενκόφσκα για την ε, καλή παρουσίαση που μας έδωσε και την προσπάθεια της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συντονίσει όλες αυτές τις πολιτικές. Πιστεύω ότι αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση για τη σημερινή μας συζήτηση. Διάβασα την ε, παρουσίασή σας με μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπω ότι δίνεται έμφαση στην βιομηχανία, ιδιαίτερα στην μεταλλουργία. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια στην ε, εξέταση και στην ε, αναθεώρηση. Υπάρχει το αρχικό στάδιο, η αναθεώρηση, ύστερα η παρουσίαση των νέων προτάσεων. Ε, μετά, να αναφερθήκατε στην βιομηχανία 4,0 και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και το πόσο, πώς μπορούμε να τη συνδέσουμε με την ψηφιοποίηση. Ε, αντίθετα από εσά, χθε το βράδυ ακούσαμε από έναν άλλο συναδελφό σα ότι σκοπεύει μέχρι το 2020 να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή αγορά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εγώ να σα ρωτήσω εάν είναι εφικτό φέτος να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την βιομηχανία 4.0 που θα καλύπτει όλους τους τομείς και τον μεγάλο όγκο δεδομένων και την ε, καινοτομία και την ψηφιοποίηση και πώς αυτό θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω πως δεν... Α, έχω λίγο χρόνο ακόμα. Ωραία. Δεν βλέπω λοιπόν, αυτή, ε, δεν βλέπω, λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την νέα εκβιομηχάνηση και για τον στόχο του 20% που ε, έχουμε διαβάσει. Πώς θα μετρηθούν αυτά τα, τα ποσοστά, αυτό το 20% πώς το έχετε υπολογίσει ή μήπω χρειάζεται νέος υπολογισμός ε, των στόχων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε δείξει εξαιρετική πειθαρχία χρονική. Κύριος Έριξον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Πιστεύω πως αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στην ε, κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα. Το πρόβλημα σήμερα στην ευρωπαϊκή οικονομία, στις ευρωπαϊκές εθνικές οικονομίες είναι ότι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Σκεφτόμαστε βράχη πρόθεσμα, ιδιαίτερα στον ε, τομέα των επενδύσεων. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στις ε, τράπεζες και στην ετόνωση των επιχειρήσεων βράχη πρόθεσμα, μια γρήγορη δηλαδή λύση. Βλέπω εδώ ότι έχουν αναλυφθεί νέες δραστηριότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, οι οποίες όμως είναι αυτό ακριβώ, είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις. Να υποθέσω ότι αυτές οι προτάσεις θα φέρουν και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα ή πώς μπορούν να συνδυαστούν με αυτούς τους ε, μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους που έχει προτείνει η Κομισιόν. Γιατί πραγματικά βλέπω ότι οι περισσότερες προτάσεις είναι βραχυπρόθεσμες και οι μακριοπρόθεσμες προτάσεις είναι η εξαίρεση. Κυρία Μπιενκόφσκα, βλέπω πως υπάρχει ένας κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαθεί σε αυτήν την βραχυπρόθεσμη προοπτική και αυτό θα είναι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Η κυρία Ένστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και από μένα, κύριε Επίτροπε, έχω τρεις ερωτήσεις για εσάς. Η πρώτη ερώτηση. Μιλήσατε για την εξέλιξη της, βιομηχ... της βιομηχανίας και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν τίθεται θέμα. Υπάρχει όμως ε, ε, μια τεράστια διαφορά ε, στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στις άλλες χώρες στην βιομηχανική εξέλιξη, στις θέσεις απασχόλησης οι οποίες λείπουν και παρατηρούνται επίσης και τεράστια ελλείμματα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις χώρες και στις άλλες χώρες όπως στην Γαλλία ή στη Γερμανία. Τι σκοπεύει λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τονώσει την βιομηχανική εξέλιξη στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έπειτα μας μιλήσατε για ένα φιλικό περιβάλλον προς τις επενδύσεις. Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ήρθε σε μια ε, κοινή ακρόαση που κάναμε και μας μίλησε και εκείνο για την ε, εξέλιξη της βιομηχανίας, για μια φιλική βιομηχανία προς τους ε, εργαζόμενους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα συνταξιδοτικά δικαιώματα, ασφαλιστικά, η φαρμακευτική ε, περίθαλψη. Και κάτι άλλο, μα είπατε ότι θέλετε να στηρίξετε την ε, αμυντική βιομηχανία και την ε, αμυντική έρευνα νέες με στρατιωτικέ στρατιωτικές τεχνικέ. Σκοπεύετε να επενδύσετε πολλά χρήματα, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα αυτό. Μπορείτε να μα αναπτύξετε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο τι ακριβώς δηλαδή προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αμυντική βιομηχανία, πώς ακριβώς, σε ποια κράτη-μέλη θα επωφεληθούν από αυτό και ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδια για αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ένστ. Ο κύριο Τζανονάτο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Καλή ανάρρωση κιόλα ε, για το μικρό πρόβλημα υγεία που έχετε. Σα ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σα παρουσία παρά το γεγονό ότι αντιμετωπίζετε ένα μικρό πρόβλημα υγεία. Θα ήθελα να επαναλάβω μια ερώτηση που έκανε και η συνάδελφο Κόμη πριν από λίγο. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό των ε, Made in, δηλαδή του άρθρου 7 του κανονισμού για την ασφάλεια. Γνωρίζετε πόσο θεωρούμε σημαντικό το γεγονός να υπάρχει ε, ένδειξη ε, προέλευσης των προϊόντων, γιατί θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο μέσο για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Δυστυχώς, ε, τον, ε, το Συμβούλιο απέριψε την ίστατη προσπάθεια συμβιβασμού και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη βούληση να γίνουν συναντήσεις σε χώρες οι οποίες είναι κατά της ε, λύσης αυτής, του Made in για να ε, προσπαθήσουν να επιλύσουν τις δυσκολίες και να βρουν και μία οδό συμβιβασμούς. Ε, κατά την άποψή μας, ο συμβιβασμός θα πρέπει να αφορά κάποιους από τους βασικούς τομείς που πρέπει να προστατεύσουμε και να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές αλλά και για τις παραγωγικές μας δραστηριότητες. Υπάρχει σίγουρα το θέμα της κλωστοβιομηχανίας ε, και των ε, κεραμικών, η κλωστοϊφαντουργία, η επίπλωση, τα κοσμήματα γνωρίζω ότι ασχολείστε με το θέμα. Θα ήθελα να μας πείτε δύο-τρία λόγια παραπάνω για το τι ακριβώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Τζενεύσκη Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Μας κάνατε μια εκτενέστατη παρουσίαση και έχω μια ερώτηση η οποία έχει σχέση με αυτά που ρώτησε και η κυρία, ε, κυρία Νίμπλερ. Έχει να κάνει με το σύστημα Κοπέρνικος και το σύστημα Γκαλιλαίο. Αυτά τα συστήματα βρίσκονται στην, ε, στο, στάδιο, στο τελικό στάδιο της θέσης σε ισχύ. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ρωτήσω τα προγράμματα αυτά, τα οποία είναι νοσιακά προγράμματα και εξαρτώνται από την συνεργασία πολλών κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς προτίθεται να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα ωφελήσει τον πολίτη ε, πώς θα ωφελήσουν μάλλον τον πολίτη αυτά τα δύο προγράμματα και πώς ε, αυτά θα ωφελήσουν και την ε, ασφάλεια θα ήθελα λοιπόν εγώ να σας ερωτήσω πώς θα χρησιμοποιηθούν, για ποιους σκοπούς τα προγράμματα αυτά. Επίσης, σε σχέση με το εμπόριο, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, τι γίνεται με τις ε, χώρε όπως η Ρωσία για παράδειγμα, με τις οποίες ε, τώρα έχουμε κάποια προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νόμιζα ότι είχα προσελκύσει την προσοχή της Γραμματείας νωρίτερα. Κυρία Επίτροπε, αναφερθήκατε στη χημική βιομηχανία ότι είναι βασικό τομέα επιτυχιών για την Ευρώπη. Τι λέτε για τα σχόλια του κύριου Jim Ratcliffe από τα μεγαλύτερα αφεντικά στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τη χημική, με τι ενεργειακέ τιμέ σημερινέ και τιμολόγηση, λέει δεν θα υπάρχει καθόλου χημική βιομηχανία ευρωπαϊκή σε 10 χρόνια. Σήμερα παρέστην σε ένα γεύμα που διοργανώθηκε από τη Χαλιβουργία. Και υπάρχουν δύο βασικέ ανησυχίε. Οι τιμέ τη ενέργεια και η υπερβολική νομοθεσία. Εξεπλάγει. Διότι σήμερα το πρωί, κυρία Επίτροπε, διάβασα την επιστολή σα και πράγματι ανταποκρίθηκα, απάντησα και το βασικό πνεύμα τη απαντήσεώ μου ήταν το εξή είπα ότι αγνοείται ή δεν δίνεται τη δέουσα προσοχή στα δύο βασικά θέματα που εμποδίζουν την βιομηχανία και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, τιμές της ενέργειας με ιονή θρησκευτική προσήλωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπερβολική ρύθμιση. Με τα χαράς βλέπω ότι στα σχόλιά σας ξεκινήσατε να ασχολείστε με το πρόβλημα των υπερβολικών ρυθμίσεων αλλά δεν βλέπω το ίδιο επίπεδο ενέργειας, ενθουσιασμού και φιλοδοξιών που απαιτείται όσον αφορά την ενέργεια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσω της ενεργειακής πολιτικής να πιέσουμε ενεργοβόρες βιομηχανίες και ε, θέσεις και επενδύσεις να φεύγουν από την Ευρώπη. Κλείνουν εγκαταστάσεις στην πετροχημικά ή βιομηχανία δηληστήρια, στη αλλουργία, τσιμέντο, τα χημικά. Όλοι φεύγουν λόγω των πολιτικών μας και πάνε σε άλλες νομοθεσίες με χαλύτερες προδιαγραφές για το περιβάλλον, όχι μόνο υπονομεύουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία του τρόπος, αλλά αυξάνουμε και τον, ε, τις εκπομπές του άνθρακος σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σύμφωνα με τους δικούς σας όρους θα έλεγα ότι θα το αποκαλούσατε τρέλα. Ευχαριστώ. Τελευταίος. Ο κ. Ουρμπαν Κρέσπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Όπως θα γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η κοινωνική οικονομία και η αλληλέγγυα οικονομία στην Ευρώπη αριθμεί 250.000 συνεταιρισμούς που απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων και έχουν ε, πάνω από 8 εκατομμύρια εταίρους πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος προσφέρει ε, προστασία της απασχόλησης και ποιότητα της απασχόλησης ενώπιον της κρίσης ε, και των μέτρων λιτότητας που η πλειονότητα των συντηρητικών αυτού του κοινοβουλίου ε, υποστήριξε και πέρασε μέτρα με την υποστήριξη και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχει δημοκρατία στην οικονομία χάρη σε εμά και υπάρχουν ε, άτομα τα οποία εξηγούν πώ πρέπει να παράγουμε ε, απλώς και μόνο για να ανταποκριθούν στι προκλήσει τη αγορά. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν κύριε Επίτροπε ποιε είναι οι συγκεκριμένε δράσεις εντός ή εκτό του προγράμματο COSME που σκοπεύετε να εφαρμόσετε για να εδραιώσουμε και να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό ιστό αυτή τη ε, αλληλέγγυα και κοινωνική οικονομία. Δεύτερον, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι περίπου το 90% των επιχειρήσεων επιχειρήσεων στη χώρα μου, στην Ισπανία και ε, είναι υπεύθυνε για το 67% της απασχόλησης ε, στην οικονομία. Παρόλα αυτά, ε, ε, το 35% κρατικές συμβάσεις. Ε, σκοπεύεται να ανοίξετε παρόλα αυτά με την DTIP, να ανοίξετε στις μεγάλες επιχειρήσεις και κοινοπραξίας να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και τελικώς να παραβιάσουν την αρχή της ελεύθερης, του ελεύθερου ανταγωνισμού με ρήτρε οι οποίες θα εισαχθούν και θα αποτελέσουν φραγμούς για το εμπόριο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής ποιες προβλέπετε εσείς ότι θα είναι οι συνέπειες ε, της TTIP ε, για τον επιχειρηματικό ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και κυρίως πώς θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει την απασχόληση ποιότητας ε, στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία ή αν αυτά μας τα λέτε αυθορμήτως. Ευχαριστώ, μακρηγορήσατε κάπως, αλλά τι να έκανα. Λυπούμε. Κυρία Επίτροπε, ήταν ο τελευταίος ε, αγορητής. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε στις τεθήσεις ερωτήσεις και τα σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα σχόλιο έχω. Σε εκείνους που δεν θα απαντήσω πλήρως ενδεχομένω ή με έναν τρόπο που θα θέλατε να σας απαντήσω, θα σας δώσω γραπτός κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, έγινε μια μελέτη που ανετέθη από μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το, βάσει 7, για το άρθρο 7 και δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο από αυτού, διότι επαναλαμβάνω αυτό που είπα στο Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά κυρίως τους συμβιβασμούς και δεν δέχομαι ότι η μισή Ευρώπη μπλοκάρει το πακέτο των αγορών, της εποπτείας των αγορών και της ασφάλειας ε, των προϊόντων λόγω ενός άρθρου που είναι σημαντικότατο για την υπόλοιπη Ευρώπη και δεν νομίζω ότι ευσταθεί αυτός αλόγος για να μπλοκάρει οι δέσμοι μέτρων. Προσπαθήσαμε να δεν έχουμε καταλήξει κάπου, δυστυχώς. διότι σύμφωνα με τη μελέτη αφορούσε τα υποδήματα και τα κεραμικά το άρθρο 7. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι κρίμα που δεν συμφωνούμε σε ένα ζήτημα ίσονος σημασίας ενώ αντιθέτως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βασικό πακέτο μέτρων για την εποπτεία των αγορών και προϊόντων, για την επαναβιομηχανοποίηση ε, μέσω μικρομεσών επιχειρήσεων. Συμφωνώ απόλυτα της κυρίας Μουμπάψκα και του κυρίου Γκέρεκ. Υπάρχει πηγή χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Έχουμε ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεως και των σχετικών εργαλείων όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το συζητώ το θέμα και με τα κράτη-μέλη πώς να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καλύτερες χρηματοδοτικές πηγές από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και από τους εθνικούς πόρους και ενιαία αγορά. Αυτό θα βοηθούσε. Το συζητούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι η ενιαία αγορά είναι κάτι που περιμένουν πώς και πώς, χωρίς κατακαιρματισμό του είδους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 28 διαφορετικά νομικά καθεστώτα και διαφορετικούς κανόνες μπορούν να ανταγωνίζονται μόνο με εξωτερικούς ανταγωνιστές αν είναι ισχυροί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι ισχυρές οι επιχειρήσεις σε μια χώρα, μέλος δεν αρκεί. Πρέπει να γίνουν ισχυρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της και μετά να συναγωνιστούν άλλους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Για βιομηχανία για όλους, να συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Πρέπει να εστιαστούμε επί υποδομών, τα μεγάλα, τα ογκώδη στοιχεία, εμπορικό εμπόριο, ε, μπλοκάρισμα υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές του κόσμου, διαχωρισμός. Έχουμε industry φυτού στην Γαλλία, industry φυράλες στη Γερμανία, έχουμε διαφορετικά προγράμματα στην Ολλανδία, στην ε, Σουηδία. Θέλουμε πανευρωπαϊκά προγράμματα δεν μπορεί μεμονωμένη κάθε χώρα να έχει δικό της πρόγραμμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ψηφιακή ενιαία αγορά. Και έχουμε και σχετικό σχέδιο δράσης. Άμυνα. Η ομάδα υψηλού επίπεδου για την έρευνα για θέματα ΚΕΠΑ συνεδρίασε άπαξ. Θα συνεδριάσει μετά το καλοκαίρι ξανά το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα ΣΕΡΠΑ εργάζεται σκληρά. Θέλουμε μέχρι το Μαρτίου του χρόνου μέσω της εκθέσεως ομάδας υψηλού επίπεδου να έχουμε εντοπίσει δύο-τρεις τεχνολογίες που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους για τρία χρόνια πριν την λήξη του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του παρόντος και μετά να χρηματοδοτηθεί η έρευνα η σχετική με την ΚΕΠΑ και η αμυντική βιομηχανία στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με ξεχωριστό κονδύλι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελείται η ομάδα από επιχειρηματίες, επιστήμονες και πολιτικούς και νομίζω ότι το κράμα είναι καλό για να εντοπίσουμε δύο, τρεις, δεν ξέρω τεχνολογίες που θα ε, χρηματοδοτηθούν από δημόσιους πόρους. Ο κύριος Έριξον είπε ότι έχουμε πολύ ε, μακροπρόθεσμες προοπτικές. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες προοπτικές, κατεπηγόντως όμως χρειαζόμαστε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα από τους πολίτες και από τη βιομηχανία και από όλους μας σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. Δεν θέλουμε ε, να το δούμε σε 20, 15, 10 χρόνια. Θέλω να έχουμε κάθε χρόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Του χρόνου, απαντώντας τον κ. Τασενόφσκι, τα λέω αυτά, του χρόνου λέω, θα έχουμε το σχέδιο δράσης για το Γαλιλαίος και πώς θα απορροφηθούν οι υπηρεσίες του από την αγορά, πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες από το Γαλιλαίος και στο τέλος για την υπερβολική νομοθεσία ρύθμιση και την ενέργεια δεν είναι κάτι που το αγνοώ. Είμαι κάθετα κατά της υπερβολικής ρύθμισης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποσυρθούν όσο το δυνατόν περισσότερες νομοθετικές προτάσεις και να πλουστεύσουμε την νομοθεσία και τους κανονισμούς όσο γίνεται. Για την ενέργεια μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν μπορούμε να είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που αυτοτραυματίζεται με πολύ ψηλού στόχους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς. Εάν όλοι κάνουν το ίδιο, καλώς. Αν η Ευρώπη όμως είναι η μόνη περιοχή του κόσμου που το κάνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί κινδύνους για την βιομηχανία μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου για τις απαντήσεις σας, για την παρουσίασή σας και ελπίζουμε ότι θα μας ξανάρθετε φέτος. Σίγουρα όχι πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές βεβαίως για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας ε, η ε, στρατηγική εξόδου από την κρίση. Να πω τώρα για τα μέλη, 15 και 16 Ιουλίου, πρωί και απόγευμα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας, επομένως θα συναντηθούμε ε, τέσσερις φορές ακόμα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, σε όλους τους υπολείπους ό,τι καλύτερο.